Μίλησα με τον Πρωθυπουργό Ράτας, ο οποίος με διαβεβαίωσε ότι το μεταναστευτικό είναι ύψης της σημασίας. Τα πρακτικά έχουν διανεμηθεί, τα πρακτικά του Ινίου υπάρχουν παρατηρήσεις, όχι, άρα εγκρίνονται.